Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Αντικαθιστώ, όπως ξέρετε, τον ε, άξιο πρόεδρό μας, τον κύριο Μπούζεκ, ο οποίος δεν μπορεί σήμερα να παρευρεθεί. Να σας παρουσιάσω τον κύριο Φεράχτατ από την Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανικών Βιοπροϊόντων και τον κύριο Βάνεμαρ Χίλτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επεξεργασία των ε, βιομηχανικών βιοπροϊόντων. Να σας θυμίσω ότι αυτή η κοινή επιχείρηση είναι η πρώτη πρωτοβουλία για τέτοιε νέε κοινέ επιχειρήσει μετά την έγκριση του Horizon 2020. Ξεκίνησε το καλοκαίρι του Υπουργέτη μετά τι επιτυχημένε διαπραγματεύσει του Ευρωκοινοβουλίου στο τέλο τη προηγούμενη θητείας και με τη συμμετοχή πολλαπλών δημόσιων και ιδιωτικών ε, εταιρικών σχέσεων. Ο κύριος Φανίστερο είναι εδώ. Τέλεια. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Είναι ο εισηγητής μας για το θέμα αυτό, σήμερα το πρωί. Και έχουμε συνολικά μία ώρα και 15 λεπτά για την παρουσίαση και τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Θα παρακαλέσω τον κύριο Φεράχτερτ να μας παρουσιάσει το όλο θέμα. Έχετε συνολικά ένα δεκάλεπτο. Thank Ευχαριστώ κύριε Henkel για την ε, παρουσίαση. Αρχικά θέλω να αποτέσω φόρο τιμή στις προσπάθειές σας στα μέλη της Επιτροπής αυτής που επέτρεψαν να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία όπως είχε προταθεί στην προηγούμενη θητεία της Επιτροπής σας. Και ιδίω, κύριε Φανίστερο, έχετε καταβάλει πολλές προσπάθειες και ήρθατε και σήμερα το πρωί πάνω απ' όλα. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια συνολική θεώρηση του τι εννοούμε από οικονομικής άποψης για την ε, ιδιωτική δημόσια αυτή εταιρική σχέση, εταιρική σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, στον τομέα των ε, βιομηχανικών βιοπροϊόντων. Και θα σας πω και τι αποτελέσματα ελπίζουμε να επιτύχουμε. Οι διαφάνειες δεν ε, εμφανίζονται ακόμα. έρχονται οι Η βιοοικονομία, κυρίες και κύριοι, βασίζεται στη χρήση των ανανεώσιμων βιολογικών <coughs> πηγών σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, κυρίως το πετρέλαιο, που είναι μη ανανεώσιμος πόρος για σκοπούς ε, χρήσης ενέργειας, για βιομηχανικούς, ε, χημικούς σκοπούς Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε στα πλαίσια της βιοοικονομίας είναι να δημιουργήσουμε ένα οικονομικό σύστημα βιωσιμότερο, ε, φιλικότερο προς το περιβάλλον, πρασινότερο και που να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στις ε, ερχόμενες γενιές. Η βιοοικονομία, λοιπόν, εξετάζει τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε καλύτερες ανανεώσιμες βιολογικές πηγές ενέργειας με βιομηχανικές διαδικασίες, αλλά και ενδεχόμενα ανοίγματα στην αγορά, για να δούμε πώς αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν. Ε, για να το πετύχουμε αυτό στην Ευρώπη, ε, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο, στη Βόρεια Αμερική στη νοτιοανατολική Ασία, σε διάφορες περιοχές της. Εκεί υπάρχουν ε, αρκετέ προσπάθειες και ιδιαίτερα ωφέλη σε σχέση με την Ευρώπη μεγαλύτερα κιόλα. Με ε, επιτυχίες στον τομέα των ε, τροφίμων και των ζωοτροφών λόγω χάρη ή με το ζαχαροκάλαμο λόγω χάρη που είναι μια πολύ φτηνή λύση για την παραγωγή δύο προϊόντων. Ε, με τα δύο δηληστήρια λόγου χάρη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί πολύ συχνά χρησιμοποιούνται σιτηρά και ε, εκεί χρησιμοποιούνται προϊόντα για βιομηχανικούς σκοπούς, αλλά μας ενδιαφέρει και η δεύτερη γενιά των καλλιεργειών που προωθούνται από τα δηληστήρια. εάν δούμε τώρα την ε, εταιρική σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, όλα αυτά γίνονται γιατί πιστεύουμε ότι παράσχεται ένα σαφέστερο πλαίσιο και για το μέλλον. Μιλάμε για μια εταιρική σχέση μεταξύ του δημόσιου τομέα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του μηχανικού κλάδου, τον ιδιωτικό. Με στήριξη από διάφορου ομίλου, λόγω χάρη στα πλαίσια του Horizon 2020. Μια από τι δυσκολίε βέβαια είναι ότι επειδή υπάρχει ένα διετή κύκλο προγραμματισμού, είναι δύσκολο να υπάρξουν μακροπόθεσμε επενδύσει επενδύσεις. Η εταιρική σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα έχει και άλλα πλέον εκτήματα, επειδή προσφέρει ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον μιας δεκαετίας. Είναι μια κοινή προσέγγιση και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε εδώ είναι να ε, οδηγήσουμε σε σύγκληση διάφορου βιομηχανικούς κλάδου, οικονομικούς φορείς που συνήθως δεν συνεργάζονται. Η εταιρική σχέση δημόσιο ιδιωτικού τομέα του προσφέρει την πλατφόρμα, προσφέρει σε αυτέ τι εταιρείε την πλατφόρμα να ενώσουν τι δυνάμεις του. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, όχι απλώς ενώνουν τις δυνάμεις τους, αλλά και τις ε, ειδικέ τους γνώσεις και τους πόρους τους. Σε δραστηριότητες που θα ήταν δύσκολο μεμονωμένα να αναπτυχθούν. Όπως με τη διοργάνωση στο PPP. Την ε, Εταιρική σχέση δηλαδή δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Επίσης έχουμε μόχλευση για μελλοντικές επενδύσεις και η χρηματοδότηση που διατίθεται για την πρωτοβουλία πρόκειται κυρίως από το Horizon 2020. Αλλά για κάθε ευρώ που διατίθεται για την πρωτοβουλία η βιομηχανία προσφέρει 2,8 από την πλευρά της ευρώ. Επίσης εξίσου σημαντικό πρόκειται για μια πρωτοβουλία στα πλαίσια του PPP, της εταιρικής αυτής σχέσης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, με ε, βασική κατεύθυνση την αγορά. Η ίδια πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δύο ε, προϊόντων. Δεν κοιτάμε λοιπόν μόνο την βιομηχανία των χημικών ή των πλαστικών ή των καυσίμων. Αλλά προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Δεν κοιτάζουμε μόνο τη δασοκομεία ή τη γεωργία. Όλα συνδυάζονται σε μια αλυσίδα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Δεν υπάρχουν αυτά ως σήμερα και οι βιομηχανικοί παράγοντες δεν τα έχουν αναπτύξει αρκετά. Λόγου χάρη, αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι με διάφορες ε, βιομηχανίε, με διάφορου μηχανικούς κλάδου, των χημικών, των καυσίμων, να πετύχουμε τη συνεργασία με τους τελικούς χρήστες. Λόγω χάρη τα καύσιμα, τα χημικά προϊόντα μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή άλλων συστατικών για τρόφιμα. Όπως είπα ξεκινώντας, η Επιτροπή σας μας στήριξε ιδιαίτερος λανσάροντας την πρωτοβουλία, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, η οποία εγκρίθηκε τελικά μέσα στο καλοκαίρι και τέθηκε επιτέλους σε ισχύ, τώρα κάνουμε τα πρώτα μας δειλά βήματα, τα πρώτα μας νηπιακά βήματα, για να το πω έτσι, στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας και σε ό,τι αφορά την αλληλοποίηση, ήδη έχουμε ξεκινήσει την πρώτη ε, διαδικασία για την υποβολή υποψηφιωτήτων και προτάσεων. Έχουμε προοικοδότηση περίπου 7 δις. Ε, τα περισσότερα έρχονται από το Horizon 2020, 2,7 δις προέρχονται από την βιομηχανία την ίδια. Ο εταίρος από την πλευρά του Δημοσίου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα είναι μια εμπορική ένωση, ε, η σύμπραξη για τα δύο προϊόντα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την πρωτοβουλία κατά την υλοποίηση του προγράμματο. Χρησιμοποιούμε του κανόνε που ισχύουν για το Horizon 2006 2020, συγγνώμη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό βάσει τη αρχή τη ανοιχτή συμμετοχή. Δηλαδή, κάθε οργανισμό ή ένωση μπορεί να συμμετάσχει βάσει των κανόνων διαφάνειας, της ανοιχτής συμμετοχής και της αριστείας. Δηλαδή, μόνο τα καλύτερα, τα βέλτιστα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν. Και όπως είπα θα επικεντρωθούμε στη δημιουργία νέων αλυσίδων παραγωγής βιοπροϊόντων με ιδιαίτερη αξία, όπως τα βιοδηληστήρια. Τώρα για τον ιδιωτικό τομέα, όπως είπαμε υπάρχει αυτή η σύμπραξη των βιο... Ε, ε, της βιομηχανίας βιοπροϊόντων με τουλάχιστον 70 μέλη, μεγάλες εταιρείες, μικρομεσές και κάποια κλάστερ. Επίσης υπάρχουν 121 συνεργαζόμενα μέλη, πανεπιστήμια, ε, ερευνητικά κέντρα και εμπορικοί οργανισμοί, καθώς και άλλοι τομεί με τι ειδικέ του γνώσει για τα χημικά, για την ενέργεια και ούτω καθεξή. Όπω θα δείτε από τη διαφάνεια, ε, μέλη έχουμε σε όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι έχει αποκλειστεί καμία ευρωπαϊκή χώρα από την όλη πρωτοβουλία, οπότε είναι πολύ αντιπροσωπευτικό ο χάρτη στο τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Έχει ξεκινήσει η πρώτη διαδικασία για την υποβολή προτάσεων ε, με η οποία θα διοργανώνεται σε αιτήσια βάση, βάση του Horizon 2020 και των κανόνων του. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο. Έληξε η όλη διαδικασία στις 15 Οκτωβρίου φέτος. Οι πρώτες προτάσεις ήδη εξετάζονται και αν όλα πάνε καλά, η πρώτη συμφωνία, ε, η πρώτη σύμβαση θα υπογραφεί το Μάρτιο φέτος. Εάν τα δούμε από μια ευρύτερη οπτική γωνία, τα θέματα της πρωτοβουλίας, βλέπουμε ότι προσπαθεί να οθήσει την ε, μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη για την Ευρώπη και την, να τονώσει επίσης την ανταγωνιστικότητά της σε μεγαλύτερη κλίμακα, δηλαδή να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη και ε, να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις από το βιομηχανικό κλάδο. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να έχουμε προγράμματα που θα επιτρέψει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, το ορυκτό πετρέλαιο δηλαδή. Θέλουμε διώσιμες ε, εναλλακτικέ εδώ, λόγω χάρη στα πλαίσια της πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές, για την ενεργειακή ασφάλεια και ούτω καθεξής για την πράσινη ανάπτυξη. Και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια. Ανέλαβε ο νέος επίτροπος για την ερεύνα και την καινοτομία, ο κύριος Μουέντας, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα ότι πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα και η πράσινη ανάπτυξη. Το είπε και στην ακρόαση στην Επιτροπή σας. Οικονομική ανάπτυξη αλλά και πράσινη. Αλλά εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη με τρόπο βιώσιμο δεν χρειάζεται καν να ασχοληθούμε. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία μας εντάσσεται πλήρως σε αυτές τις προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φεράχτερτ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συντονιστές και θα αρχίσουμε με τον κύριο Βανίστελ Ρόι, ο οποίος είναι και ο πρώην εισηγητής της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι πλέον μέλος της Επιτροπής Ήτρε, αλλά θα παρακολουθήσω το θέμα σε κάθε του στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ε, γρήγορη αρχή και εφαρμογή του προγράμματος, διότι σε πολλά προγράμματα και στον ορίζοντα 2020 παρατηρούμε καθυστερήσεις. Υπάρχουν πολύ απλήρωτοι λογαριασμοί, όμως αυτή είναι μια νέα πρωτοβουλία και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδιστεί από τα υπολείμματα της προηγούμενης περίοδου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας συγχαρώ για το μεγάλο ενδιαφέρον που έχετε δείξει. Έπειτα, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι όλες οι χώρες θα συμμετέχουν σε αυτήν την νέα πρωτοβουλία και όλες οι περιφέρειες και όλα τα πανεπιστήμια και όλες οι επιχειρήσεις λοιπόν από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πάρα πολύ καλό διότι στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020 είδαμε ότι το 90% των προγραμμάτων αυτών είχαν εφαρμοστεί στα παλιά κράτη-μέλη. Και η δύο οικονομία είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να ωφελήσει ιδιαίτερα χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και άλλες. Και πραγματικά βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον από αυτές τις νέες χώρες οι οποίες δεν εκπροσωπούνται στους, στους ομίλους και στις ε, συμπράξεις μέχρι τώρα. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σχόλιο σχετικά με το τι συμβαίνει στα προγράμματα αυτά. Η έξυπνη εξειδίκευση. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βιοοικονομία και αυτές οι πρωτοβουλίες θα εφαρμοστούν σε περιοχές ε, όπως ε, περιοχές της Πολωνίας, στο Λουμπλίν για παράδειγμα. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι ακόμα τελειοποιημένα, όμως είναι πολύ χρήσιμο είναι πολύ χρήσιμα για τις περιοχές αυτές και πραγματικά πρέπει να τις προσέξουμε, διότι μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικές για αυτές τις περιοχές τώρα, όμως θα είναι σε λίγα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτήν την πολύ γρήγορη αρχή του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νίστελ για τη συνεισφορά σας στο θέμα αυτό. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόπες Περμέγιο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε αυτό ο υποτομέα τη βιομηχανία επέκτησε προτεραιότητα όσον αφορά τις ε, επενδύσεις του δυτικού τομέα και αυτό πρόκειται να δώσει ε, σε ένα τομέα έντασης κεφαλαίου ιδιαίτερη όθηση και αυτό γιατί εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε να έχουμε στα θέσεις εργασία και ε, θα πρέπει βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με τις ΜΜΕ που την χάνουν οι κρατικών επιδοτήσεων. Πάντως ακριβώς εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί φραγμοί ούτως ώστε να μπει κάποιος καινούριο στην αγορά και αυτό λόγω του ότι χρειάζονται πάρα πολύ σημαντικές ε, επενδύσεις για το υλικό, για τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Οπότε ε, επ' αυτού θέλω να σας ρωτήσω τι μέτρα ε, σύμπραξη δημόσιο ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να γίνουν τόσο ώστε να μπορέσουμε ακριβώ να άρουμε αυτά τα, αυτούς τους φραγμούς της ε, πρόσβασης για τις ε, ΜΜΕ και τέτοιου είδους ε, χρηματοδότηση ε, σημαίνει βοήθεια στις μεγάλες εταιρείε που δεν έχουν περιορισμούς κεφαλαίου αλλά αυτό ισχύει σαν φραγμός για τις ΜΜΕ. Τι, τι θα γίνει με το με το, με το, με το για να αποτιμητήσουμε αυτή ε, ε, αυτόν τον περιορισμό. Οπότε, οπότε τώρα θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ε, αντίστοιχη ρύθμιση των στόχων των επιχειρήσεων και κάποια συστήματα ελέγχου, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτά τα προγράμματα. Εάν το συνδέσουμε σε άλλους εμπλεκόμενους της ΜΜΕ και από την άλλη μεριά να έχουμε μόνο ωφέλεια των μεγάλων εταιριών, αυτό το πρόγραμμα τότε γίνεται μια φάρσα, γίνεται ένα δεκανίκι για τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Σας ερωτώ, τι μηχανισμούς αξιολόγησης έχουμε τόσο ώστε να ξέρουμε τον υπολογισμό των ΜΜΕ, άμεση στήριξη και τι είδους ωφέλειες και που προκύψουν για αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριε Γκρίφιν, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να κάνω ένα παρόμοιο σχολείο με το δικό σας σχετικά με το REACH. Η βιοβιομηχανία και η βιοοικονομία είναι πάρα πολύ σημαντική στις ε, περιοχές της υπαίθρου σε όλο το τμήμα τη βόρεια Αγγλία. και παρατήρησα στο χάρτη που μα δείξατε ότι οι κοινοπραξίε αυτέ δεν συμπεριλαμβάνουν τη Βόρεια Αγγλία, το Βόρειο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια που κάνουν πραγματικά καινοτόμα δουλειά εκεί. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώ θα προσεγγίσετε αυτές ε, αυτά τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια στην Βόρεια Αγγλία για να συμμετέχουν και εκείνα σε εκείνη την πραγματικά σημαντική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να η περιοχή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αγνώστ. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα αυτό και είναι γνωστό αυτό. αυτό που είναι πιο σημαντικό όμως είναι να συμμετέχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ε, τομέα αυτό. Και για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθούν κλάστερ ανάμεσα στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές και τα πανεπιστήμια. Να δημιουργηθούν συνεργασίες έτσι ώστε να δημιουργηθούν με τη σειρά τους θέσεις απασχόλησης. σε αυτό το project συγκεκριμένα υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες όπου να παρατηρείται συνεργασία ανάμεσα σε πανεπιστήμια και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν ναι, πώς προωθούνται αυτές οι συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βιλκόναν έχει το λόγο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό αυτές οι εταιρείες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγαλύτερες να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους από όλη την Ευρώπη σε συνεργασία με πανεπιστήμια και τις αρχές τοπικής Είναι ένα πολύ καλό μήνυμα και είναι σημαντικό η ανάπτυξη νέων προϊόντων να λάβει την απαραίτητη σημασία. Ιδίω για τα δευτερεγέννη προϊόντα, για τα παράγωγα από τη γεωργία, τη δασοκομεία. Ωστόσο, έχω και μία απορία. Δεν θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε στην νομοθεσία να μην υπάρχουν φραγμοί για να μπορεί κανείς να αντλήσει ωφέλη από αυτά τα νέα προϊόντα και να συνεχίσει όλη αυτή η προσπάθεια. Δεν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις κατάλληλες πρώτες για να παράγουμε ενέργεια. Γνωρίζετε εάν υπάρχει κάποιο νομοθέτημα, κάποια νομοθετική πράξη που να αποτελεί φραγμό, για σε αυτή την περίπτωση που οπωσδήποτε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χάμνερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην παρουσίαση υπήρχε μία φράση η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον ότι το project δηλαδή αυτό δημιουργεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ε, όπως γνωρίζετε υπάρχει μια συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα βιοκαύσιμα, με την έμεση αλλαγή χρήσης της γης και με όλα αυτά τα θέματα. Αλλά ένα πράγμα που δεν έχουμε δει ακόμα στην ε, όλη ιστορία με τα βιοκαύσιμα είναι αυτές οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ε, το αντίθετο μάλιστα έχουμε δει ε, περίπτωση όπου τα ευρωπαϊκά όργανα δημιουργούν προϋποθέσεις στις οποίες η βιομηχανία θα επενδύσει πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά και μετά ε, έχει δεύτερη σκέψη για τα βιοκαύσιμα, για τη χρήση τους και ύστερα αλλάζουν οι κανόνες. Αυτό υπονομεύει εντελώς αυτές τις επενδύσεις ε, στις οποίες αναφερθήκατε και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτά τα προγράμματα που συζητούμε εδώ θα είναι, θα επηρεαστούν από αυτήν την αλλαγή, ακριβώς όπως επηρεάστηκαν και τα βιοκαύσιμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χέλμερ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτήν την πρωτοβουλία και την εφαρμογή της. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, διότι γνωρίζουμε όλοι πόσο χρειάζεται να ε, προωθηθεί και να ενισχυθεί ε, ο χώρος των βιοκαυσίμων. Φυσικά χρειάζεται να γίνουν οι προτάσεις, να ελεγχθούν αυτές οι προτάσεις και έπειτα να προχωρήσουμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς συνεργάζεστε με τα κρατημέλη. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ίδρυμα το οποίο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των προγραμμάτων του Ορίζοντα 2020. Συνεργάζεστε λοιπόν εσείς με αυτές τις επιχειρήσεις και τα ίδρυματα έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τις συνεργασίες αυτές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάπελ. Άλλε ερωτήσει. Όχι από ό,τι βλέπω. Έχετε πέντε λεπτά τώρα για να απαντήσετε όλες μαζί τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Um, try and take ε, the questions in order. Για να δούμε τις ερωτήσεις. Άκουσα τι είπε ο κ. Φανίτσελβάη όσον αφορά τα περιφερειακά ταμεία, την εξειδίκευση. Και συμφωνώ μαζί σας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την πρωτοβουλία μας. Δεν μπορούμε να έχουμε βιοοικονομία ευρωπαϊκή εάν δεν έχουμε βιοοικονομίες ε, τοπικές και περιφερειακές. Σας το λέω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Αλλά με στην παλαιά οικονομία είχαμε την βιομηχανία σε μια βιοοικονομία, έχουμε την ε, βιοοικονομία η οποία έρχεται στην, ε, στις ζωοτροφές, στο δάσος, όπου, όπου χρειάζεται. Ναι, είναι αναπόφευκτο να έχουμε τέτοιες συνέργειες που θα πρόκειται να δημιουργηθούν τώρα. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι παραδεχόμαστε ότι είναι κλειδί για την επιτυχία της πρωτοβουλίας μας η ΜΜΕ. Λάβαμε μια σειρά μέτρων για να εξασφαλίσουμε ότι οι ΜΜΕ θα έχουν τη θέση που τους αξίζει. Στο κονσόρτσιουμ αυτό έχουμε φορείς που εκπροσωπούν ΜΜΕ και με μεμονωμένες ΜΜΕ και κάθονται γύρω από το τραπέζι καθώς συζητούμε το του προγράμματος. Ευθύς εξ αρχής αυτής της διαδρομής. και είπαμε να εξασφαλίσουμε το πώ, όσον αφορά την έρευνα θα έχουμε χρηματοδότηση για τι ΜΜΕ. Φόρειο ερευνητική, πανεπιστήμια, να είναι επιλέξιμε οι ΜΜΕ για χρηματοδότηση. To financial resources available under the initiative. And of course, uh, Επίσης, όπως και για το Horizon 2020, η ΜΜΕ πρόκειται να είναι επιλέξιμες για τον στόχο που έχουμε τάξει για αυτό το 20% που προβλέπει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία. Οπότε και θεωρούμε ότι με αυτά τα μέτρα που έχουμε λάβει οι ΜΜΕ θα συμμετάσχουν. Βεβαίως θα υπάρχει εποπτεία προσεκτική και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Τώρα σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο νομίζω ότι υπήρξε κάποια περιμηνία των όσων είπαμε. Είπαμε συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Δεν είπαμε ότι μόνο ο Νότος θα εκπροσωπηθεί. So I'll try and make it to, to, to, to ensure that this uh, yellow circle is in the middle and not, uh, not at the bottom there. Είδατε, είδατε το, το σχετικό σημάδι, αυτός ο, το κίτρινο σημάδι και ο κίτρινο κύκλος είναι στη μέση της χώρας, δεν είναι κάτω-κάτω, στον νότο. Οπότε πρέπει να εμπλέξουμε τις ε, περιφέρειες. Μόνο έτσι θα πετύχει η πρωτοβουλία μας. Άρα συμμετέχει και το Βόρειο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, σε σχέση με τους φραγμούς νομοθετικής φύσεως. Και αυτό είναι βέβαια πολύ σημαντικό και σίγουρα δεν αρκεί. Να έχουμε δράσεις για να δεν προβλέπονται τα μέτρα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν την αγορά καθεαυτή. αυτή. Άρα κοιτούμε θέματα σαν την τυποποίηση, κάποιες πιστοποιήσεις, ε, κάποιες διατάξεις για τις κρατικές προμήθειες. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς επιτροπής για την βιομηχανία. Και έτσι έχουμε νοτήσει δραστηριότητα, ούτως ώστε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις ευθύς εξ αρχής. Τώρα, κάποιος αναφέρθηκε στα βιοκαύσιμα. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε υπόψη μας, οπωσδήποτε. Είναι σωστή πρωτοβουλία αυτή. Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρξει εκτροπή. Γιατί αν αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίσουμε, τότε μπορεί να πάρουν στραβή, άσχημη τροπή τα πράγματα. Καταναλωτές, ρυθμιστικές αρχές, αγορά, όλες αυτές τις μεταβλητές τις λαμβάνουν υπόψη. Και θέλουμε από την αρχή να εμπλέκονται όλοι αυτοί. Μην έχουμε τελικά μόνο τα νέα προϊόντα τα οποία να προωθούμε και αυτά να μην ενδιαφέρουν τον κόσμο. Επίσης, όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, όσον αφορά την διακυβέρνηση, έχουμε την ομάδα εκπροσώπων των κρατών. Υπάρχονται συμβουλές και εκεί, στη φάση ανάπτυξης της πρωτοβουλίας, εμπλέκονται τα κράτη-μέλη. Και έχει να κάνει αυτό και με την περιφερειακή διάσταση. Τα κράτη-μέλη έχουν αποφασιστικό ρόλο στο πώ θα μπει στην αγορά αυτή η πρωτοβουλία. Κύριε Φεράφτερ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ ο και σα ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ να έρθετε και να μα παρουσιάσετε την εισήγησή σα και να, να απαντήσετε τι ερωτήσει. Και σα ευχαριστούμε κύριε. Uh, ladies and gentlemen, <clears throat> let us now approach the second subject of this morning, which is... Uh, το δεύτερο θέμα της ε, σημερινής συνεδρίας, που είναι το Horizon 2020, ε, τεχνολογίες ε, κλειδί, όθηση για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία ή στον κατασκευαστικό ή μεταποιητικό τομέα. Έχουμε και εδώ μια σύγχυση και ετοιμάστε και τις δικές σας ερωτήσεις στη συνέχεια. Οπότε τώρα θα σας παρουσιάσουμε τον κύριο Χόφερτ Χέσπερς και τον κύριο Μπέτερ από το TNO. TNO είναι η ο Ολλανδικός Φορέας για τις εφαρμοσμένες επιστήμες. Καλώς ορίσατε κύριε. Εσείς είστε ο κύριος Χέσπερς. Καλώς ορίσατε. Yes, okay. Oh. Mr. Okay. You get some help, no? <clears throat> So, uh, <clears throat> ladies and gentlemen, this study which uh, is requested by the... Έχουμε αυτή την μελέτη, την οποία την ζήτησε και την παρήγγειλε η Επιτροπή μας. Για αυτές τις τεχνολογίες κλειδί. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για την βιομηχανία κατασκευαστική, μεταποιητική. Οπότε τώρα παρακαλώ, ο κ. Χέσπερς μπορεί τώρα να μας κάνει την εισήγησή του για αυτήν την μελέτη. Έχετε 10 λεπτά κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μας χαρά να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης. Μας δώσατε μόνο 10 λεπτά, οπότε και θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχαίως. Πρώτα-πρώτα να σας πούμε τις αδρές γραμμές της εισήγησής μας κατόπιν της έκθεσης και μετά να σας πούμε τα βασικότερα σημεία. Πρώτα πρώτα είπαμε ποιες είναι αυτές οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τώρα να δούμε το, το πλαίσιο αυτών των στόχων. Η Ευρώπη βγαίνει από μια σοβαρή κρίση και οικονομική ύφεση, αλλά χρειαζόμαστε νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης, ούτω ώστε να δυναμώσουμε, να δώσουμε και ενούργια ζωτικότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Και οπότε βασικός στόχος εδώ είναι <clears throat> η πρωτοπορία σε αυτές τις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Έχουμε μια ανακοίνωση και δύο ομάδες υψηλού επίπεδου για αυτές τις τεχνολογίες. Έξι τέτοιες τεχνολογίες μας απασχόλησαν και θα επανέλθουμε σε αυτό. Και αυτά τα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια του Οριζόντου αλλά και σε άλλα προγράμματα. στόχο τη μελέτη είναι να μπορέσουν τα μέλη τη επιτροπή σα να διαμορφώσουν την απόψή του για το πώ αυτέ οι τεχνολογίε βοηθούν την έρευνα, την καινοτομία και την βιομηχανία και βέβαια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δύο λόγια τώρα για αυτές τις τεχνολογίες, μια που δεν έχουμε τον χρόνο να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες. Νανοτεχνολογία, νανοηλεκτρονική, ημιαγωγή, προωθημένα υλικά, βιοτεχνολογία, βιομηχανική, που συζητήσατε πριν από λίγο, προχωρημένα συστήματα μεταποιητικά, κατασκευαστικά. Μία συν πέντε έξι τέτοιες τεχνολογίες λοιπόν, γνώση, έρευνα και ανάπτυξη που από ένταση και εργατικό δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων. Απαιτούνται δαπάνες ε, αρκετά ευξημένες για τα καινοτόμα νέα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. Είναι συστημική σημασία σε αυτό για τα θεμέλια της βιομηχανίας. Για να τα δούμε τώρα στο ευρύτερο παγκόσμιο πιο σφαιρικό πλαίσιο είναι πρωτοπόρα η Ευρώπη όσον αφορά τη δημιουργία γνώσης και για τις ευρεσιτεχνίες, δημοσιεύσεις, όμως χάνουμε έδαφος σε σχέση με τους ε, ανταγωνιστές όσον αφορά την εκμετάλλευση αυτής της ε, γνώσης. Και αυτό οφείλεται στην κοιλάδα του θανάτου στα σχετικά προγράμματα. Είδαμε τι γίνεται με την Ασία Όμως η Ασία χάνει κάπως εδαφός γιατί το εργατικό κόστος στην Κίνα αυξάνεται. Και η ρομποτική επίσης έχει συρρυκνώσει την σημασία της εργατικής δύναμης όσον αφορά το κατασκευαστικό μεταπητικό τομέα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με ε, αυτές τις ε, ομάδες Γκρενόμπλ, Γερμανία, η κοιλάδα βιολογική Δανία κλπ. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις κοιλάδες του θανάτου, τις επωνομαζόμενες. Είναι μία έννοια η οποία έχει εισαχθεί για να χαρακτηρίσουμε το πώς οι τεχνολογίες οδηγούν σε προϊόντα. Άρα χρειαζόμαστε εδώ τρεις πυλώνες για να γεφυρώσουμε αυτήν την κοινότητα. τεχνολογικό, πρωτότυπο και ανταγωνιστική κατασκευή, ούτως ώστε αυτά η, η, τεχνολογίες να αποκτήσουν κάποια συγκεκριμένη αξία. Και δεν είναι μόνο τεχνολογική η κοιλάδα του θανάτου. Γι' αυτό και σε κάποιες μελέτες επισημαίνονται δύο διαφορετικές κοιλάδες. Μία τεχνολογική και μία σε σχέση με τη θέση σε εμπορία, την καινοτομία και τα επιχειρηματικά μοντέλα. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ούτε τη μία ούτε την άλλη μορφή. δούμε τώρα το επίπεδο ενάργειας αυτής της τεχνολογίας. Πρωτότυπα, ε, επιχειρηματικότητα και, και τέλος πάντων διάφορα στάδια και οδηγούν στην κατασκευή του προϊόντος, στην παραγωγή. Έχουμε επομένως αυτά τα εννέα βήματα, τα βλεπω κατω κάτω-κάτω σε αυτή τη διαφάνεια. το επίπεδο και τη ετοιμότητα τέλο πάντων τη τεχνολογία, πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε πάνω πάνω στην, ε, ε, στη διαφάνεια αυτή. Άρχισαν νέα μοντέλα επιχειρηματικά για να τώρα να επιταχύνουμε όπω πιέζει ο χρόνο για να δούμε τώρα πώ γίνεται να έχουμε μια αποτελεσματική στατική όσον αφορά αυτέ τι τεχνολογίε. Βλέπουμε εδώ πέρα ε, με πηγή το κάτινα τη ε, Γενική Διεύθυνση για τι Επιχειρήσει. Έχουμε εδώ πέρα την προσαρμογή των οργάνων, των μέσων και των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε κάποιε δομέ διακυβέρνηση και επίση χρειαζόμαστε και κάποιο είδου εμπορικά μέσα πολιτική, ώστε να υπάρχει και στον αγωνισμό. Πάμε τώρα στην επόμενη. Διαφάνεια. Τι γίνεται σχέση με το ορίζον 2020. Δεν γίνεται σχέση με άλλε ενωσιακέ δραστηριότητες και μέσα πολιτικές. Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε μια προϋποδότηση 30 δι για το ορίζον 2020. Η προτεραιότητα δίνεται σε κάποια πιλωτικά στοιχεία, ούτως ώστε τα πρωτότυπα να γίνουν ε, ε γίνουν προϊόντα ε, μέσω της παραγωγής αυτών. Όμως, Αυτές, αυτά τα πιλωτικά στοιχεία και η θέση εμπορία προϋποθέτουν ε, ετοιμότητα τεχνολογική υψηλό επίπεδο. Το θέμα βέβαια είναι τώρα κάποιοι κανόνες, κάποιες διατάξεις κρατικής ενίσχυσης. Αυτό δεν είναι πάντα ένα πρόβλημα, ε, είναι προβληματικό στη φάση της παραγωγής. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει σημαντική συμμετοχή της βιομηχανίας και θα πρέπει η κυβέρνηση να φροντίζει να μην έχουμε στρέβλωση της αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε υποδομές. Θα πρέπει σχετικές διευκολύνσεις να χρησιμοποιούνται από περισσότερους χρήστες και επίσης το θέμα είναι σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι πρωτοπόρα η βιομηχανία που είναι κοντά στην αγορά και αυτές οι τεχνολογίες έχουν να κάνουν με στρατηγική έρευνα, με καινοτομία και με την ε, ε, είσοδο των προϊόντων στην αγορά. Τώρα πιο συγκεκριμένα έχουμε τον πρώτο πυλώνα 13 δις ERC FET. Δεύτερος πυλώνας 17 ε, δις βιομηχανική πρωτοπορία και εδώ έχουμε και τις τεχνολογίες ε, καινοτομία ΜΜΕ, επίσης έχουμε τις κοινωνικές προκλήσεις. Εδώ δεν έχουμε συγκεκριμένη πληκοδότηση, αλλά έχουμε υποστήριξη για την καινοτομία. Επίσης έχουμε ε, εταιρική σχέση για το Horizon 2020, για, τα, για το KIC και το Evrica, Δράσεις του Horizon 2020. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχουμε και θέματα πέραν του 2020, του ορίου του 2020, στατηγικές εξειδίκευσης, να δούμε τι γίνεται με τις ε, τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Ε, ο ρόλος οικονομικών μέσων πολιτικής που θα αφορούν και το 2020 και άλλα προγράμματα. Να ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την χρηματοδότηση, την ΜΕΝ με την ΔΕ. Το 2020 δηλαδή, το 2020, με τους διαρθρωτικούς πόρους για να αποφύγουμε παντός είδους επικάλυψη. Επιταχύνω γιατί πιέζει ο χρόνος. Και κλείνουμε ρίχνοντας μία ματιά για το τι γίνεται όσον αφορά τις δεξιότητες, την απασχόληση κλπ. Νέες τεχνολογίες. Βιομηχανία που βασίζεται στις ε, τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Σχεδιασμός προϊόντων, έρευνα, ανάπτυξη, όλα αυτά έχουν εδώ να παίξουν το ρόλο τους πολύ σημαντικά. Να προσέξουμε τις νέες δεξιότητες. Επίσης το θέμα είναι ότι αν έχουμε κάποιο είδους κενό, χάσμα εδώ όσον αφορά τις δεξιότητες των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. Η απάντηση είναι καταφατική. Έχουμε τώρα άλλες δύο διαφάνειες. Επικεντρώνουμε στο πόδι με αυτές τις ε, τεχνολογίες σε έξι επιμέρους από αυτές. Χρειάζεται η ευελιξία όσον αφορά την επιλογή, γιατί αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Ας πούμε το λογισμικό ε, είναι και τομέα όπου εδώ πέρα λείπει η παρουσία της, γενικής, της τεχνολογίας γενικής εφαρμογής. Είναι και το θέμα της τεχνολογικής όθησης, συμμετοχή επίσης των ΜΜΕ για να πετύχουμε το στόχο της βιομηχανικής πρωτοπορίας οι υποδομές που αφορούν περισσότερους χρήστες, το είπαμε αυτό πριν, συνδυασμός χρηματοδότησης και πόρων, και αυτό εδώ πέρα έχει κάποια θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά επίσης και η αποτελεσματική χρήση και ανάπτυξη τεχνολογιών ε, για επιχειρηματικά μοντέλα, έρευνες, τελευταία τώρα διαφάνεια, ο συνδυασμός του ορίζουν 2020 για των ιδιωτικών ταμείων είναι πάρα πολύ βασικό, τόσο ώστε να φτάσουμε στην κρίσιμη μάζα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επένδυση. Αλλά εδώ πέρα έχουμε τους στόχους που είναι για το ορίζον 2002 η αριστεία και για τα διορθωτικά ταμεία της ε, μη ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αναφέραμε την ορισμένη προσέγγιση ώστε να καλύψουμε όλη την αλυσίδα της ε, αυτή την αλυσίδα της διαδρομής αυτής, value chain και επίσης εδώ να δούμε το ότι ανάντι και κατάντι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες και θα χρειαστούν επομένως, θα χρειαστεί η ανάπτυξη ιδιαίτερα ε, προχωρημένων δεξιοτήτων. Ευχαριστούμε κύριε Ισπέρης. Ε, πραγματικά νομίζω το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μελετήσετε αυτό το τόσο ενδιαφέρον έγγραφο. Είναι μια εξαιρετική μελέτη του όλου θέματος. Να περάσουμε τώρα στους συντονιστές. Και πάλι έχουμε τον κύριο Φανίστερ ο οποίος ε, έχει παρακολουθήσει το, όλη, το όλο εγχείρημα με μεγάλη προσοχή. Ναι, μιλήσαμε ήδη για την βιοοικονομία και σχετίζεται άμεσα και με το θέμα που τώρα συζητάμε. Κατά πρώτον, είναι πολύ καλές αυτές οι επιλογές, αλλά υπάρχει και άλλη μία ερώτηση. Δηλαδή, ε, εδώ ε, προβλέπουμε 20 δις. Θέλουμε να υπάρξει παραγωγή καλής τεχνολογίας, αλλά μετά θα την πουλήσουμε στην Ασία. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα δίνουμε κονδύλια θα εκπαιδεύουμε ανθρώπους και μετά θα τα πουλάμε αλλού. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες όπως από την Ολλανδία ή άλλες ε, πολυεθνικές, η Samsung, αυτοί αναγκάστηκαν να έρθουν στην Ευρώπη όταν δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Εάν δεν προστατεύσουμε τις γνώσεις μας και κάτι ακόμη δεν περιλαμβάνεται στο φυλάδιο για τις κρατικές ε, βοήθειες. Το Horizon 2020 είναι σε πιλωτική φάση. Μπορούμε να πάμε παραπέρα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήδη το κάνουν στο πιλωτικό rollout Κάνουν πολύ περισσότερα. Μπορούμε λοιπόν να μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς να το ρισκάρουμε για αργότερα. Και ε, τρίτον, η σχέση με τα διευθυντικά ταμεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δαπανούμε 20% και έχουμε ανανεώσει τους στόχους αυτής της πολιτικής ε, για το 2020 λέγοντας ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η γνώση και η καινοτομία. Πρώτη προτεραιότητα είναι οι υποδομές γνώσης, είναι η εκπαίδευση των πολιτών. Σωστά λοιπόν το είπατε, και το σχολιάσατε ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους συμμετέχοντες και για, τα, για όσους συμμετέχουν στα ΚΕΤ και για τα πανεπιστήμια και για τα εθνικά κράτη. Υπάρχουν λοιπόν εδώ διαφορετικοί κανόνες, μπορούν να αξιοποιηθούν, αλλά πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο. Ε, αυτή τη στιγμή ε, σε άλλο σημείο της, ε, των Βρυξελών γίνεται μια μεγάλη διάσκεψη για τα ΚΕΤΣ. Νομίζω ότι κι άλλοι θα τα σχολιάσουν αυτά, όπως και εγώ και θα συμφωνήσουν μαζί μου. Ευχαριστούμε. Κυρία, Κυρία ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στη σύνδεση ανάμεσα στον ορίζοντα 2020 και την πολιτική συνοχής. Πολύ σωστά είπατε ότι ο ορίζοντας 2020 θέλει να προωθήσει την αριστεία και η πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη των περιφερειών. Όμως, όταν βλέπω πόσα κονδύλια διατίθενται στην ε, πολιτική συνοχή και δεδομένου ότι η έρευνα και η ανάπτυξη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτική συνοχής και να πω και ότι προέρχομαι από μια περιοχή από την Σαξονία η οποία έχει τρομερές ελλειψει όσον αφορά την πρόθεση ανάπτυξης αναρωτιέμαι τι κάνουμε στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 έτσι ώστε να συνδυάσουμε όλα αυτά με την ε, διαρθρωτική πολιτική και αν κάνουμε αρκετά πράγματα έτσι ώστε πραγματικά ο συνδυασμός των ε, δύο αυτών ε, πολιτικών να επιφέρει αποτελέσματα. Μιλάμε για έξυπνη πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιες προϋποθέσεις δημιουργούμε έτσι ώστε να την χρησιμοποιήσουμε διότι Πράγματι παρατηρούνται ελλείψεις ε, όσον αφορά τη σύνδεσή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τεμποράνο. Μία ερώτηση σε σχέση με τις ε, τεχνολογίες για την εκτύπωση την τρισδιάστατη. Μπορεί αυτή η τεχνολογική διαδικασία να θεωρηθεί και έτσι. και τι κονδύλια θα χρειάζονταν για ανάπτυξη σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών στα προγράμματα ορίζοντα 2020. Αυτές οι καθυστερήσεις έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που είπε και η συνάδελφος για την συνένωση του ορίζοντα 2020 με, την, ε, με τα διαθερωτικά ταμεία, ε, θα ήθελα να εστιάσω καταρχάς και στο Μάντσεστερ, τη δική μου περιφέρεια, αλλά θα ήθελα να πω ότι πρέπει και οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ε, θέσεις απασχόλησης έτσι ώστε και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης υψηλέ θέσει απασχόληση στι περιφέρειε αυτέ. Πώ μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όλα αυτά τα προγράμματα θα ε, συνδυαστούν έτσι ώστε να δημιουργηθούν υψηλού επίπεδου θέσει απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρίφιν. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δεν βλέπω να ζητήσω ζητά κάποιος το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στους εισηγητές για να απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Όσον αφορά λοιπόν τις μεγάλες επενδύσεις και εάν θα χάσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εάν θα μας ξεπεράσει η Ασία και πώς να προστατεύσουμε τις γνώσεις μας και την καινοτομία μας. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τα μέσα που έχουμε. Υπάρχουν κάποια παραδοσιακά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όμως από την μελέτη μας προέκυψε ότι εάν επιταχυνθεί ο ρυθμός της καινοτομίας, αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην αλυσίδα αξιών και στο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας. Θα είμαστε λοιπόν πολύ ταχύτεροι στη μετάβαση από βασικές τεχνολογίες και την ανάπτυξη αυτών σε παραγωγή πρωτότυπης και καινοτομάς τεχνολογίας. Πιστεύω πως αυτό είναι βασικό έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πρωτοπορία. διότι πραγματικά ο διεθνής ανταγωνισμός θα αυξηθεί. Και για να διατηρηθούμε στο προσκήνιο πρέπει να μάθουμε από τις εμπειρίες μας, να διδαχθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να καινοτομήσουμε ταχύτερα και πώς μπορούμε να είμαστε ταχύτεροι στην επεξεργασία των ε, προϊόντων και στην εφαρμογή των ε, νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτό θα είναι και η καλύτερη εγγύηση για την Ευρώπη έτσι ώστε στο μέλλον να παραμείνει σε ηγετική θέση. Όσο για τη δεύτερη ερώτηση, ο συνάδελφός μου θα απαντήσει σε αυτή. Επιτρέψτε μου και εμένα να πω δύο λόγια για την πρώτη ερώτηση. Ε, έχει συζητηθεί πολύ το θέμα πολλές δαπάνες, μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα και μετά τα αποτελέσματα να φεύγουν και να διαφεύγουν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ένα φαινόμενο υπερχείλησης, για να το πούμε έτσι, spillover. Εάν ε, λοιπόν γίνουν τέτοιες επενδύσεις στην Ευρώπη, σίγουρα σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές, λόγω της έρευνα και ανάπτυξης, θα υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο μετάδοσης. Ε, αλλά και στις δικές μας τις περιοχές. Το σημαντικό εδώ είναι ότι το R&D, η έρευνα και ανάπτυξη, είναι μια παγκόσμια ε, προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η έρευνα θα γίνεται στην Ευρώπη και μετά θα μένει μόνο στην Ευρώπη για να την εξυπηρετεί. Εάν το απαιτούσαμε αυτό, θα χάναμε τις διασυνδέσεις με άλλες περιοχές του κόσμου και είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά ένα από τα πορίσματα της ε, μελέτης είναι ότι πρέπει να κοιτάξει κανείς τι γίνεται και στη συνέχεια ε, της ε, όλης προσπάθειας. Δηλαδή τι γίνεται στην Ευρώπη για να αξιοποιηθεί όλη αυτή η έρευνα. Πολλοί, ε, όπως η SML, παίρνουν πολύ καλή χρηματοδότηση από τη Samsung, από άλλες εταιρείες, αλλά αυτή αυτά τα κονδύλια, αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να κατευθυνθεί στι μικρέ περιοχέ τη Ευρώπη, στι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση και στι περιφέρειε, για να υπάρξει περαιτέρω τόνωση τη έρευνα. Έπειτα για την ε, διαφυγή τη παραγωγή προ τι ΗΠΑ. Πολλά γίνονται στι ΗΠΑ, αλλά πιο πολύ ακόμη στην Ασία. Και προσπαθούν να αποσπάσουν όσα περισσότερα μπορούν από την έρευνα. Όμως θα το καταλάβετε και από το πρόγραμμα που κάναμε για τα πολλαπλά ΚΕΤ για τις Ηνωμένε Πολιτείες και είδαμε ότι από το πρότυπο προϊόν μέχρι το πιλωτικό και τη μαζική παραγωγή, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Στο ομοσπονδιακό τουλάχιστον επίπεδο. Όμως σε επίπεδο πολιτιών μπορεί να χρηματοδοτείται λόγου χάρη ε, κάτι πολύ συγκεκριμένο, ε, όπως η φούντι. Αλλά... Αλλά Αυτά είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με την Ευρώπη. Και νομίζουμε ότι συνδυασμός με το Horizon 2020 μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Οι τέσσερις ελευταίες ερωτήσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και αν το, η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι και. Η απάντηση είναι ναι, είναι. Είναι πολύ περίπλοκη η τεχνολογική μέθοδος έχει να κάνει και με την κατασκευή αλλά και με τη μικροκενάνο ηλεκτρονική. Χρειάζονται υψηλότατες δεξιότητες. Ε, είναι εντατική και η χρήση κεφαλαίων. Όλα τα κουτάκια συμπληρώνονται για να θεωρηθεί και έτσι. Ναι, και τις άλλες δύο ερωτήσεις. Για την, για την ερώτηση του συσχετισμού μεταξύ του Horizon 2020 και του Ταμείου Συνοχής, αν αυτός ο συσχετισμός, αν αυτή η σύνδεση είναι αρκετά ισχυρή και αν τα αξιοποιούμε καταλήλως, η απάντηση θα πρέπει να είναι νομίζω όχι ακόμα. Έχουμε αναφέρει κάποιες από τις ε, δυσκολίες που υπόκεινται. που υπάρχουν εδώ. Το Horizon 2020 προωθεί την αριστεία και την καινοτομία. Στη συνοχή υπάρχει άλλη λογική. Δεν είναι εύκολο πάντοτε να υπάρχει σωστή διασύνδεση. Όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ολοκληρωμένη αλυσίδα καινοτομία από την έρευνα και το πιλωτικό στάδιο στην μεταποιητική βιομηχανία. Η συμμετοχή των διαφορετικών ταμείων σε αυτή την προσπάθεια στήριξη για την βιομηχανία κατασκευή και με στρατηγικέ εξειδικευσεί μπορεί να αντιμετωπίσουν και προβλήματα. Αυτό όμω που είναι σίγουρα απαραίτητο είναι να έχουμε κάποια πειραματική δράση, κάποια εργαστήρια, κάποιες διαδικασίες που επιτρέπουν να διδαχθούμε από τον συνδυασμό αυτών των δύο διαφορετικών προγραμμάτων, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το Horizon θα προωθεί την αριστεία και ε, την καινοτομία και τα διευθυντικά ταμεία θα παίρνουν τον μπαλάκι και θα το πετάνε στο επόμενο γήπεδο τη μεταπητική βιομηχανία. Αλλά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για να πετύχει αυτό. Και τελευταία ερώτηση. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. πολύ ισχυρό δεσμό μεταξύ διαθετικών ταμείων και Horizon 2020, διότι χρειαζόμαστε δεξιότητε. Και αν λέμε ότι χρειαζόμαστε δεξιότητε για τα ΚΕΤ, χρειαζόμαστε και μηχανικού και διδακτορικού και εργατικό δυναμικό με ιδιαίτερε δυνατότητε. Δηλαδή αυτού που μπορούν να χειριστούν και να τα βγάλουν πέρα με τα ρομπότ και τα εργαλεία προηγμένης τεχνολογία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι όλοι από τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνία. Μπορεί να είναι και εργάτες, εργαζόμενοι που ε, έρχονται από εργοστάσια. Και εκεί χρειάζεται κάποια επένδυση. Σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη των ΚΕΤ με τη γυρά του πληθυσμού στην Ευρώπη και τη συνταξιοδότηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού την ερχόμενη δεκαετία, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να αναβαθμίσουμε τις επενδύσεις μας στις δεξιότητες για να παραμείνουμε στη διεθνή προσκήνιο πρωταγωνιστές. Ευχαριστούμε. Εφόσον υπήρξατε τόσο πειθαρχημένοι, ίσως για το δεύτερο θέμα να βιάστηκα και να μην έδωσα χρόνο για ερωτήσεις. Κύριε Ετσενίκε, και μετά ο κύριος Φανίστερο για δεύτερη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Η φωτονική, η νοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία. Είναι τέτοιες τεχνολογίε γενική εφαρμογές όπως αυτές που είπε συζητούμε, αλλά επίσης αυτό το οποίο ισχύει είναι το ότι η κοινωνική τεχνολογία είναι κάτι πάρα πολύ βασικό και είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. το πιο σημαντικό κομμάτι της επιστήμης αλλά και της τεχνολογίας είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω και σας ερωτώ τι μέτρα σχεδιάζετε να λάβετε ούτως ώστε να σταθεροποιήσετε, να εξασφαλίσετε τους ερευνητές μας γιατί πολλές φορές η σταδιοδρομία τους χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια απίστευτη επαγγελματική. Και πολλές από τις οικογένειές τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μια ακόμη ερώτηση για την έρευνα. Το τι βάζουμε στην έρευνα και τι παίρνουμε. Μιλάμε για ένα παγκοσμιοποιημένο τοπίο, για ροές αλλά πώς βλέπετε να εξελίσσονται τεχνολογικές λύσεις για νέες μπαταρίες. Από ό,τι ξέρω δεν παράγουμε πλέον μπαταρίες στην Ευρώπη. Δεν αρκεί να λέμε ότι ε, ότι όλα αυτά τα ε, έχει πάρει η και κάνει ό,τι θέλει. πρέπει να δούμε εμείς πώς θα χαράξουμε τη βιομηχανική μας πολιτική. Οι εταιρείε μπορούν να πουλάνε ό,τι θέλουν. Άμα θέλουν μπορούν και να ξεπουλήσουν. Τώρα βλέπουμε να, να έχει γεράσει ένα μέρος του πληθυσμού. Σε λίγα χρόνια θα έχουμε ακόμα περισσότερους. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τη γνώση για την παραγωγικότητα στην Ευρώπη. Ίσως υπήρξαμε πολύ απλόχεροι. Πολύ εύκολα τη χαρίσαμε τη γνώση μας. Έτσι μας λέτε εσείς λειτουργούν τα πράγματα και υπάρχουν και καλά παραδείγματα αλλά εγώ ανησυχώ λιγάκι. Ίσως να μην ε, βρίσκεται αυτό το πεδίο της μελέτης σας αλλά πρέπει να το σχολιάσω. Πρόεδρος, έχω ακόμη δύο συμμετέχοντες και μετά θα έλεγα να σταματήσουμε. Κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τονίσατε στην αρχή της ομιλίας σας πόσο σημαντική είναι η καινοτομία και η κατασκευή στον ε, τομέα αυτό. Τι γίνεται για να προωθηθούν αυτή οι τομείς έτσι ώστε να αποφύγουμε να πέσουμε σε αυτήν την κοιλάδα του θανάτου που αναφέρατε. Ε, επίσης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και η διάθεση στην αγορά, ο τρίτος τομέας και αυτός ο τομέας είναι ε, ένας τομέας που έχει πάρα πολύ καλό δυναμικό όμως υπάρχουν πάρα πολύ λίγα ε, μέσα για να τον προωθήσουμε. Τι μπορείτε να κάνετε για να αναπληρωθεί το κενό αυτό, να αναπληρωθούν αυτές οι ελλείψεις που έχουμε όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά αυτών των ε, τεχνολογιών. Έχουμε δηλαδή αυτά τα πολύ καινοτόμα προϊόντα και τι τεχνολογίε που δημιουργούνται στην Ευρώπη, δεν διατίθενται όμω στην ευρωπαϊκή αγορά επειδή λείπουν οι δυνατότητε. Γι' αυτό λοιπόν ε, η ερώτησή μου είναι, υπάρχουν προβλέψει για δημιουργία τέτοιων μέσων τόνωση τη ε, διάθεση στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κουντίσκα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι δεν συμφωνώ με την ε, αποτίμηση της έκθεσής σας. Ιδίω αυτό που αναφέρεται στη σελίδα 67 στα συμπεράσματα. Εκεί λέει η έκθεση ότι εάν στηρίξουμε προγράμματα μέσω των διευθυντικών ταμείων ιδίως στις ε, μειονεκτούσες περιοχές, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην είναι αρκετά τα κονδύλια και να μην καλυφθούν οι περιοχές που είναι ήδη προηγμένες. Νομίζω ότι πάει λίγο μακριά το συμπερασμά σας, διότι πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της έρευνας και των ακαδημαϊκών ε, γνώσεων βρίσκεται στο επίπεδο των περιφερειών, ιδίως στα νέα κράτη-μέλη, που έχουν ήδη επενδύσει σε εργαστήρια και ανάλογες υποδομές. Στο προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στην Πολωνία η κυβέρνηση είχε στόχο να φροντίσει να υπάρξουν επενδύσεις στα εργαστήρια και την, ε, τις υποδομές εχμής. Νομίζω το ίδιο ισχύει και σε άλλες χώρες. Εφόσον λοιπόν έχουμε τέτοιου είδους εργαστήρια, φροντίσουμε να έχουμε και τη βασική συνεργασία που χρειάζεται από όλους τους ε, έχοντες την, ε, τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό στη διάθεσή τους για τον σκοπό των ΚΕΤΣ. Νομίζω οι μειονεκτούσες περιοχές μπορούν να αναπτυχθούν αρκετά γρήγορα, διότι μπορούν να ακολουθήσουν το δρόμο της εξειδίκευσης. Μπορεί να γίνουν βασικά κέντρα, κι κέντρα και να προσελκύσουν ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Και τώρα τελευταία ερώτηση από τον κύριο Ζωρίνιου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το θέμα το βασικό που τέθηκε εδώ είναι το πώς θα διατηρήσουμε στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μεγάλο μέρος της ε, προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από αυτές τις ε, τεχνολογίες. Και εδώ υπάρχουν δύο σοβαρά σχόλια. Ένα είναι η ο σχηματισμός σε κλάστερ. Θα πρέπει να προβλέψουμε 4-5 διεθνή κλάστερ που να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Ευρώπη και να αξιοποιούνται και αυτές τις τεχνολογίες. Δηλαδή να βρεθούν σε αυτό το πλαίσιο των κλάστερ των σχηματισμών που θα ε, ε, εμποδίσουν την ε, διαφυγή των γνώσεων αυτών, των τεχνολογιών προς την Ασία. Κάτι που θα έπλετε τη δική μας απασχόληση. Για κάτι ακόμη που αφορά τις ε, περισσότερες χώρες μας. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που στηρίζονται από ε, δημόσια κονδύλια που γρήγορα πολλούνται και πολύ γρήγορα φεύγουν από τα χέρια μας. Σημαντικό είναι λοιπόν να έχουμε δημόσιους πόρους ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ώστε τα διπλώματα αυτά που έχουν που έχουν προκύψει από τα δημόσια κονδύλια να δημιουργήσουν μια τέτοια κρίσιμη μάζα ώστε να προστατεύουμε τη γνώση που αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Okay, thank you very much. Ευχαριστούμε. Κύριε Χίσπερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, η οποία απαιτεί, αποτελεί συνέχεια τη προηγούμενη για του ανθρώπινου πόρου. και το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα κέτς. Όντω. για τις βασικές τεχνολογικές γενικές εφαρμογές είναι πολύ σημαντική. Οι άνθρωποι και οι ανθρώπινοι πόροι. Όμω υπάρχουν σοβαρέ διαφορέ μεταξύ των διαφορών, ευρωπαϊκών χωρών. Σε πολλέ χώρε άνθρωποι με υψηλά προσόντα δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Δεν του απορροφά ο κλάδος τη βιομηχανία. Ενώ υπάρχουν άλλε χώρε. βασίζονται σε Ινδούς και Κινέζους μηχανικούς <coughs> Εάν δείτε τι γίνεται σε πολλά από τα τεχνικά μας ιδρύματα, ένα μεγάλο ποσοστό μάλιστα των φοιτητών, ε, ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών είναι φιάτες. Εάν υπάρχουν τάσεις αλλαγής σε όλη, την Ευρώπη, δεν το ξέρω, αλλά θετικά μηνύματα έχουμε από διάφορες χώρες. Όπως με την αύξηση των ενδιαφέροντό ε, ε, για τη μηχανική. Τα πολυτεχνία, τα μαθηματικά, τις επιστήμες, τις θετικές επιστήμες, διότι ακριβώς επιτρέπουν να βρει κανείς δουλειά σε ένα υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας, της ε, βιομηχανίας. Τα πανεπιστήμια προέβλεψαν θέσεις για νέους φοιτητές Σε μερικές χώρες λοιπόν ισχύει αυτό, ενώ σε άλλες η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Εδώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω πολλά μπορούν να γίνουν προκειμένου να υπάρξουν θέσεις εργασίας για ανθρώπους με ψηλά προσόντα και από χώρες που ταλανίζονται από την ανεργία των νέων. Νομίζω εδώ έχουμε πολλά να κάνουμε. Ο συνάδελφος θα απαντήσει στο δεύτερο σημείο. Yes, that's, uh, the, continuous, uh, Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν. Παίρνω τη σκητάλη από τον κύριο Φανίστελ Ρόι. Ε, αναφερθήκατε στο πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης και στις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και τις διαρροές προς άλλες περιοχές του κόσμου. Πιστεύω πως οι μεγάλες εταιρείες είναι πολύ σημαντικές. Είναι κόμβοι για την Ευρώπη. Αλλά όχι για την ε, δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Οι μεγάλες αυτές εταιρείες, το αντίθετο μάλιστα, έχουν όλο και λιγότερες ε, θέσεις απασχόλησης, διότι μέσω της αυτοματοποίησης υπάρχουν άλλοι ε, τρόποι για εξοικονόμηση κόστους. Γίνεται Γίνονται μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Και το σημαντικό είναι ότι αυτές οι εταιρείες δίνουν μεγάλη όθηση σε αυτή και προωθούν την έρευνα και την ανάπτυξη. Στην Ευρώπη πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό είναι το σημαντικότερο. και η δημιουργία βασικών τεχνολογιών εφαρμογής από τις μεγάλες εταιρείες είναι φυσικά πολύ σημαντική για την κατάντη συσχέτιση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Infineon. Η Infineon δημιουργεί στην Αυστρία ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας και έχει τη δυνατότητα να δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα προϊόντα τους έτσι ώστε να τα επεξεργαστούν. Βλέπουμε λοιπόν την δημιουργία ενός συστήματος που καλύπτει όλη την αλυσίδα αξιών. Η λύση λοιπόν δεν είναι να προλάβουμε τις διαρροές της δικής μας έρευνας και ανάπτυξης σε άλλες περιοχές. Πιστεύω πως πρέπει αντίθετα να είμαστε προορατικοί έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι και οι μεγαλύτερες εταιρείε θα έχουν ένα δίκτυο μικρότερων επιχειρήσεων γιατί αυτό είναι σημαντικό για αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό θα δώσει την αναγκαία τόνωση για να ενισχυθεί η παρουσία του στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπήρχαν και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Λέει ο κύριος Κέισπαρς. Έγινε μία ερώτηση για τη σύνδεση του ορίζοντα 2020 με τα διαρθρωτικά ταμεία. και για το πώς θα υποφεληθούν ορισμένες περιφέρειες από αυτή τη σύνδεση. Πιστεύω πως το παράδειγμα της Πολωνίας είναι χαρακτηριστικό. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια για τη δημιουργία δυνατοτήτων και αυτό είναι πραγματικά ό,τι χρειάζεται στις περιφέρειες αυτές. Υπάρχουν και άλλες περιφέρειες στις οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα επενδύσεις σε τεχνολογικές δυνατότητες και εδώ υπάρχει η δυνατότητα να αναλυφθεί πρωτοβουλία από αυτές τις περιφέρειες και να δημιουργηθεί βάση για περαιτέρω εκβιομηχάνηση και στον κατασκευαστικό τομέα. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα των περιφερειών και την ανάπτυξη των περιφερειών. Και θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις ε, νέες ε, αναπτυσσόμενες περιφέρειες και στις ε, ήδη ανεπτυγμένες. Φυσικά και υπάρχουν διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια. Ενδεχομένω υπάρχουν νέε περιφέρειε οι οποίε έχουν μεγαλύτερο δυναμικό και κάποιε οι οποίε έχουν μικρότερο δυναμικό. Υπάρχουν ορισμένε ε, ήδη αναπτυγμένε περιφέρειε οι οποίε ε, αντιμετωπίζουν μεταβατικά προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η σύνδεση του ορίζοντα 2020 με τα αρθρωτικά ταμεία, αλλά πρέπει να βλέπουμε ξεχωριστά την κάθε μία περιφέρεια, τις ειδικέ της ιδιαιτερότητες και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά για να δράσουν συμπληρωματικά. Κάθε περιφέρεια λοιπόν χρειάζεται διαφορετική στρατηγική και αυτό είναι και το σκεπτικό της έξυπνης εξειδίκευσης, ότι δηλαδή αναπτύσσεις τις δικές σου ιδιαιτερότητες. Έγινε και μια ερώτηση για το μάρκετινγκ. Υπάρχουν πιλωτικές γραμμές και πιλωτικά σχέδια και το marketing είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτών. Πρέπει να δούμε πώς θα διατεθούν τα προϊόντα αυτά στην αγορά και αυτό θα γίνει με το marketing. Και στην παρουσίασή μας αναφερθήκαμε στο marketing των προϊόντων, αλλά πρέπει να δούμε και την περαιτέρω οργάνωση της διάθεσης στην αγορά, να δούμε και την περαιτέρω δημιουργία αγοράς. Πράγματι υπάρχει περιορισμένη έμφαση στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 όσον αφορά την ε, στήριξη του μάρκετινγκ. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με την παρατήρησή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Και θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι χθες το βράδυ έγινε η συνεδρία των συντονιστών. Πρώτα πρώτα απεφάσισαν να ανατεθούν οι εξή οικονομοδοτήσει μήνων του χαρακτήρα από τα πρώτα το θέμα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τη χρήση των πόρων, κάτι το οποίο αφορούσε του ε, πρασίνου, γιατί τώρα το θέμα ε, θα γίνει κάτι το οποίο θα καλύψει αυτή την κυκλική οικονομία και επίσης από την ΚΟΕ σώμα την οικονομική, κοινωνική, εδαφική συνοχή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ρωτώ, κάτι για τα διάφορα. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Θα σα πω από την επόμενη συνεδρίαση. Στι 17 Νοεμβρίου. 3 με 6.30 στις Βρυξέλλες. Καλή σας μέρα.